Να ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις. Έχω λάβει από τους σοσιαλιστές ε, το αίτημα ο κ. Τζοβάνι Μπαρμπακάλου να οριστεί μέλος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και μέλος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες Μασρέκ. Παρατηρήσεις υπάρχουν, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν οι ορισμοί αυτοί. Να δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Τάρανς. Παρακαλώ. Un peu de silence, s'il vous plaît. Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Ε, merci, Madame Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική στον και προσωπία ε, στα θεωρία μητέρες, πατέρες της δημοκρατίας. Παρακαλώ να τους καλωσορίσουν στα θεωρία.